αριθμός ε, ε, ευρωβουλευτών που αριθμούν το, ε, στο κατώτατο κατέφλι μπορούν να ζητήσουν μέχρι την 3η 4 Απριλίου αύριο στις, στα μεσάνυχτα να επικυρωθεί απόφαση μέσω ψηφοφορίας. Εάν δεν υπάρξει τέτοιο αίτημα μπορούν να ξεκινήσουν οι αρμόδιες επιτροπές στις διαπραγματεύσεις. Να ενημερώσω επίσης ότι την Τετάρτη